On va alors commencer. Ας ξεκινήσουμε, αν είστε όλοι έτοιμοι. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα και στον ε, δόκτωρα Μουκουέγγε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir. Είναι μεγάλη τιμή που μπορώ να σας υποδεχθώ σήμερα μαζί με τους συναδέλφους Ανδρέη Πλένκοβιτς, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων, Μωρίς Πόγκα, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και, του και μαζί με τον κύριο Λουί Μισελ, Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για τις σχέσεις Ευρω... Ε, ΑΚΕ... ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν τυχόν δεν γνωρίζετε τον δόκτορα Μουκουέγγε, σας παρουσιάζω τον άνθρωπο που φροντίζει τις γυναίκες που θεραπεύει τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι η πιο απλή και σαφής περιγραφή της προσωπικότητάς του. Τον καλωσορίζουμε θερμά σε μια δύσκολη βραδιά. Σήμερα εδώ στο Στρασβούργο βλέπω ότι έχουμε αρκετές απουσίες με σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Κάποιοι συνάδελφοι ξέρω ότι έχουν μείνει στο δρόμο κάπου ε, θα έρθουν αργότερα. Ο κύριος Μικουέγγι όμως θα είναι μαζί μας ως και την Τετάρτη, οπότε θα έχουμε το χρόνο να τον συναντήσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Τιμάται φέτος λοιπόν με το βραβείο Ζαχάροφ, είναι γυναικολόγος, ε, γιατρός ε, στην, στο νοσοκομείο Πάντσι, στο Νότιο Κονγκό. Είναι εκείνος που μας υπενθυμίζει ότι έχει μετατραπεί σε όπλο μασικής καταστροφής, ο βιασμός. Έχει καταστρέψει ήδη πολλές κοινότητες, γυναίκες και οικογένειες, χωριά. Και ελπίζω ότι η βοήθεια αυτού του διάπειρου αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μας βοηθήσει να απαλείψουμε αυτά τα προβλήματα για το μέλλον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια βιώσιμη και η φόρο ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον ε, Ντένις Μουκουέγκε, θα συνομιλήσουμε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία ήταν η ζωή του, η πορεία του, η εξειδίκευσή του, οι δυσκολίες επίσης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, πολύ άριθμες δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες. Δίνω το λόγο στον κύριο Πόγκα τώρα, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και μετά στον κύριο Πλένκοβιτ, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο κύριο Μουκουέγκε και εν τέλει ο κύριο Λουί Μισελ. Και μετά θα δώσουμε χρόνο ομιλία στου συναδέλφου που τον έχουν ζητήσει και όσων ζητούν από εδώ και πάνω. Κύριε Πόγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ε, δόκτωρα Μουκβέγκε, είναι μεγάλη τιμή ως πρώτος αντιπρόεδρος ε, της ε, τροπής ε, Ανάπτυξης να σας τιμήσουμε εδώ και να σας δεχτούμε σήμερα. Γνωρίζουμε τη στράτευσή σας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας και ιδιαίτερα στο χειρουργικό σας έργο φροντίζοντας γυναίκες οι οποίες έχουν ακροτηριαστεί, έχουν βιαστεί κλπ τους ε, δίνεται την αξιοπρέπειά τους, το πνεύμα τους, την ελπίδα τους. Ε, το έργο σας είναι εξαιρετικό. Η στράτευσή σας όμως ε, δεν σταματά εκεί. Αγωνίζεστε υπέρ της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερο για την ελευθερία έκφρασης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αλλά και πιο γενικότερα, πιο ευρύτερα στην, λίμνη των, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών και ακόμα πιο πέρα. Ε, είστε στρατευμένος λοιπόν ε, και γι' αυτό το λόγο επιλεχθήκατε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τιμηθήκατε με το βραβείο Ζαχάροφ 2014. Το αξίζετε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλο σας το έργο. Ε, επισκευάζετε τις ψυχές και τα σώματα πολυάριθμων θυμάτων ε, στην περιοχή σας ο βιασμός και η χρήση του ως όπλου σε πολεμικές ζώνες και σε περιοχές σύραξης ε, είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί και να καταγγελθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας τη στράτευση και το κουράγιο σας. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Πλένκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλενθιάνο, Μαρτίνε Ορόσκο, αγαπητέ κύριε Μακουέγκε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και συμπροεδρεύω τη σημερινή συνεδρίασης. Ο κύριο Έλμαρ Μπροκ, πρόεδρο Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μα. Από το 1998 δίνουμε το βραβείο Ζαχάροβ για την ελευθερία τη σκέψη σε ανθρώπου ή οργανώσει που μέσω τη δράση του, μέσω των μαρτυριών του, μα υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι για τη δημοκρατική ζωή μια χώρα να σεβαζόμαστε και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Με την πάροδο του χρόνου το βραβείο αυτό έχει γίνει μία από τις πιο σαφείς εκφράσεις, μπορούμε να πούμε, της συλλογική μας δέσμευσης για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υποστήριξή μας προς ανθρώπους εκείνους οι οποίοι σε καθημερινή βάση μάχονται για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη παντού στον κόσμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στον κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι και πολλές ομάδες συνεχίζουν και δουν τη μάχη αυτή για τα θεμελιώδη δικαιώματα προκειμένου να καταφέρουν να καθορίσουν καλύτερα τη δική τους ζωή και το δικό τους το μέλλον φέτος και για να πω εκ νέου πάλι συγχαρητήρια στον γιατρό Μακουέκε. Το βραβείο δόθηκε λοιπόν στον κύριο Μακουέκε και η διάσκεψη των Προέδρων Αναγνώρισε επίσης τον αγώνα του Μαϊντάνα στην Ουκρανία, καθώς επίσης και τον αγώνα της Λέιλα Γιούνους ως σημαντικότατη ακτιβίστρια στο Αρζεμπαϊτζάν. Στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα προς τους ε, ανθρώπους ε, που βρίσκονται στα αντολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πραγματικά υποστηρίζουμε τον αγώνα που δίνουν για την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ενημερώθηκα ότι η εκπρόσωπη του κ. Μαντέν θα είναι στην τελετή απονομή ε, του βραβείου Ζαχάροφ την Τετάρτη. Δυστυχώ όμω η κυρία Γιούνου εξακολουθεί και βρίσκεται στη φυλακή. Η υγεία τη επιδεινώνεται και μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ακόμα για το Αρζεμπαϊτζάν. Παρ' όλα αυτά, η Τινάρα Γιούνους, η κόρη τη, θα είναι παρούσα στην τελετή απονομή του βραβείου Ζαχάροφ και θα μπορέσει να πάρει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τιμούμε σήμερα τον βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ τον γιατρό Ντένι Μακουέγγε και τιμούμε παράλληλα όλους εκείνους τους ανθρώπους που σε καθημερινή βάση δίνουν έναν σημαντικότατο αγώνα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ολοκληρώνω αναφερόμενο σε κάτι που είπε η Έλενα Ρούσβελτ κατά την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκινούν σε κάποια μικρά μέρη, κοντά στις χώρες μας, κοντά στα σπίτια μας. Τόσο μικρά τελικά μέρη τα οποία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε σε κανένα χάρτη του κόσμου. Ξεκινάνε λοιπόν στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα γρόκτημα, σε ένα γραφείο. Σε μέρη μηδαμινά όπου α, οι άντρε, οι γυναίκε, τα παιδιά αναζητούν ίσε ευκαιρίε, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια ισότιμη, χωρί καμία διακριτική μεταχείριση. Χωρί κάποια συλλογική δράση για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα μικρά αυτά μέρη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία πρόοδο στον ευρύτερο κόσμο. Σα ευχαριστώ πολύ. Απόψε έρχομαι με μεγάλη συγκίνηση αλλά και μεγάλη ελπίδα σε αυτή την πρώτη συνάντηση με τους ευρωβουλευτές. Θα ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προεδρεύει, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον Αντιπρόεδρο επίσης της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων για τη συμμετοχή τους. Θα ευχαριστήσω και τον κύριο Λουί Μισελ για την παρουσία του απόψε εδώ. με βαθιά ευγνωμοσύνη. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο έχει γνωρίσει την πιο ζωφερή περίοδο της ιστορίας της. Με 20 χρόνια πολέμων, πολέμου που δεν ακολούθησε δυστυχώς τις κλασικές, τον κλασικό τύπο και μορφή του πολέμου. Ενός πολέμου που αναπτύχθηκε εις βάρος του σώματος των γυναικών. Και βρεθήκαμε σε συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μας, σε μια περιοχή όπου βλέπαμε να διεξακόνται τραγωδίες. Το 1999 και ενώ είχαμε ιδρύσει το, νοσοκομείο του Πάντζη για να βοηθήσουμε ε, κυρίως ε, να βελτιώσουμε τους όρους της ε, περιγενετικής, ε, της μεταγενετικής μάλλον θνησιμότητας των βρεφών που είναι πολύ ψηλή στην περιοχή αυτή. Διαπιστώσαμε ένα νέο φαινόμενο, μια νέα παθολογία. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι ήταν ε, τυχαίο, συμπτωματικό ή και περιστασιακό φαινόμενο. Δυστυχώς όμως, την πρώτη αυτή χρονιά, το 1999, χρειάστηκε να φροντίσουμε 45 θύματα βιασμών με ακραία χρησιβίας. Και πρέπει εδώ να κάνουμε μια διάκριση εξάπαντος. Ανάμεσα στο βιασμό που είναι μη συνενετική σεξουαλική σχέση, που ήδη είναι ένα βαρύτατο γεγονός γιατί έχει συνέπειες για το θύμα που μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή αλλά πρέπει να τον διακρίνουμε από τον βιασμό που χρησιμοποιείται ως όπλο στον πόλεμο που όχι μόνο αφαιρεί την ανθρωπιά, ταπεινώνει, ατιμάζει και προσπαθεί ταυτόχρονα και να καταστρέψει την ε, πύλη εισόδου στη ζωή. Και πρέπει να πω ότι είναι ένας τρόπος να απαρνούνται, να απαρνηθεί την ανθρωπιά στη γυναίκα, αν δει κανείς τι συμβαίνει πάνω στο σώμα της. Το σώμα αυτό που είναι φορέα ζωής. Τα φροντίσαμε λοιπόν τα θέματα αυτά και ένα χρόνο μετά αντιληφθήκαμε ότι ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί απλώς και μόνο σε μια παράπλευρη συνέπεια ενός πολέμου. Διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συνέβαιναν αυτοί οι βιασμοί ήταν δραστηριότητες προγραμματισμένες. Δεν είναι δυνατόν σε ένα χωριό να πέσουν θύματα βιασμού μέσα σε μια βραδιά 200 γυναίκες χωρίς αυτό να έχει προγραμματιστεί προηγουμένως. Και επίσης παρατηρήσαμε στο σώμα των γυναίκων, στα σώματα των γυναικών ότι οι βιασμοί αυτοί έφεραν υπογραφή των βιαστών. Μπορούσαμε ακόμη και να διακρίνουμε με ευχέρεια τις αμοιχές, τα τραύματα ανάλογα με το σε ποια ομάδα ανήκαν οι βιαστές και αρχίσαμε να διερωτόμαστε για τους βιασμούς αυτούς στην περιοχή. Έχουμε μέχρι τώρα φροντίσει 42.000 γυναίκες που επέσαν από τέτοιου είδους σεξουαλική βία. Τις ε, φροντίζουμε με ένα ολιστικό μοντέλο. Αρχικά είχαμε επικεντρωθεί στην σωματική θεραπεία, την ιατρική φροντίδα μόνο. Διαπιστώσαμε όμως πολύ γρήγορα ότι η, η ζημία ψυχολογική ήταν τόσο βαθιά που δεν επέτρεπε στη γυναίκα να ξαναγυρίσει σε μια φυσιολογική ζωή. Και έτσι φροντίσαμε να, έχουμε, να δώσουμε και ψυχολογική υποστήριξη στις δύσκολες συνθήκες που γνωρίζει η περιοχή μας. Και σιγά σιγά δώσαμε και τη δυνατότητα για νομική αρρωγή διότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη ζωή μιας γυναίκας χρειάζεται και η απόδοση δικαιοσύνης και η αναγνώριση ότι δεν υπήρξε αυτή η υποστήριξη. Και άρα χρειάζεται η αναγνώριση και η αποκατάσταση. Και ακόμα και αν περάσει κανείς τα τρία αυτά στάδια χρειάζεται να προσφερθεί υποστήριξη και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της γυναίκας. Γιατί όταν οι γυναίκες είναι ισχυρές οικονομικά μπορούν να επαναταχθούν στην κοινωνία. Όχι γιατί θέλει η κοινωνία να τις αποδεχθεί, αλλά γιατί ξέρουν τι μπορούν να κάνουν και έχουν την τεχνογνωσία. Είχαμε κάποια πρότυπα επιτυχημένα που η γυναίκα μπόρεσε να προσφέρει κάτι περισσότερο στην κοινωνία και αυτό συνέβη όταν η κοινωνία στράφηκε προς τη γυναίκα και όχι η γυναίκα έψαξε να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία. Με την τραγωδία αυτή λοιπόν προσπαθήσαμε ταυτόχρονα να έρθουμε σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παντού, να αφυπνίσουμε την ε, διεθνή κοινότητα. Δυστυχώς όμως βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια εκοφαντική σιωπή απέναντι στο φαινόμενο αυτό το πρόβλημα αυτό που δεν είναι, θα το υπογραμμίσω, πρόβλημα των γυναικών, είναι πρόβλημα ανθρωπιάς και ανθρωπότητας. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να απομονώσουμε λέγοντας μια ομάδα και μπορεί να ρυθμιστεί από αυτή την ομάδα. Όχι, είναι κάτι που πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Και έτσι αρχίσαμε να ζητούμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε, να δώσουμε την ενημέρωση και να καταγγείλουμε ώστε να σταματήσει πια να χρησιμοποιείται ο βιασμός ως όπλο στον πόλεμο. Ο λαός του Κονγκό τώρα διψάει για ειρήνη και ανάπτυξη. Ύστερα από 20 χρόνια πολέμου, 20 χρόνια χωρίς ειρήνη και ενώ έχουμε υπογράψει πολυάριθμες συνθήκες ειρήνης, όλες αυτές οι συνθήκες είχαν δυστυχώς επαναληπτικά ένα... είχαν μέσα τους τη ρίζα της επανάληψης. Είχαμε τη συμφωνία της Αντισαμπέπα η οποία είναι για μας μια ε, συμφωνία ειρήνης και ελπίδας γιατί είναι η πρώτη η οποία δεν ενέχει, εμπεριέχει τη ρίζα της επανάληψης της σύγκρουσης στην περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ήθελα να δώσω μόνο τον τόνο αυτού που θα ήθελα να συζητηθεί σήμερα. να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια παρακολούθηση, μια συνοδεία σε αυτή την πορεία προς την ειρήνη και την ανάπτυξη για αυτό το κράτος, για αυτή τη χώρα που έχει καταστραφεί από τους πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μας υποστηρίζει πάρα πολύ. Με το βραβείο αυτό, το βραβείο Ζαχάροφ, βλέπω ότι ο λαός ε, στο Κονγκό, στην Ανατολή ή στη δύση της χώρας δεν έχει σημασία, γιατί εγώ απέχω χιλιόμετρα από την Κινσάσα, αλλά ε, το μήνυμα περνάει παρόλα αυτά ότι δεν έχουμε λησμονηθεί, ότι δεν είμαστε καταλελειμμένοι. Θα έχουμε λοιπόν τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για να μας βοηθήσει, αυτό ζητάμε, να μας βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πολιτική και διπλωματική δέσμευση το 2013, άνευ προηγουμένου, που γέννησε την ελπίδα σε όλους ότι το πρόβλημα πια μπορεί να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εμφανιστεί ως εγκύτρια αυτής της ε, Συμφωνίας Ειρήνης όπως και άλλοι εταίροι που δεν θέλω να απαριθμίσω. Το 2014 όμως σήμερα διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται ε, εμπόδια στην υλοποίηση αυτής της ε, συμφωνίας γιατί το χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί όχι μόνο καθυστέρησε λόγω της διαπραγμάτευσης Καμπάλα αλλά και ταυτόχρονα γιατί διαπιστώνουμε ότι οι συμφωνίες δεν προχωρούν όπως τα θέλαμε στην περιοχή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα παίρνει κανείς αν κοιτάξει μόνο την κατάσταση στην ασφάλεια, στη δημόσια ασφάλεια στην Ανατολή, στη Δύση της χώρας που επιδεινώνεται διαρκώς. Καθημερινά μας έρχονται πληροφορίες για σφαγές και βιασμούς που είναι μεν λιγότεροι μεν, αλλά αλλάζουν ως στρατηγική τη μορφή τους και πια ο κόσμος ανησυχεί και αδειμονεί. Γίνονται διαδηλώσεις, γυναίκες οι οποίες δεν ανέχονται πια να βλέπουν ε, να παρακολουθούν τους βιασμούς των ε, κοριτσιών τους. Έχουμε περιοχές που εκδηλώνονται σφαγές, ανησυχητικά δηλαδή δείγματα. Και νομίζω ότι το να μιλούμε σήμερα για λύση, για να αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία και άρα να καταπολεμηθούν οι βιοπρεγές αυτές που αναπτύσσονται σε περιβάλλον εμπόλεμο, σημαίνει ταυτόχρονα και ενίσχυση του αγώνα για κατά της ατιμορρησίας, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι γυναίκες αυτές που έχουν βιαστεί και περιμένουμε ακόμα μέχρι και σήμερα τη δικαιοσύνη πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με τους δημίους τους οι γυναίκες αυτές, δημίους οι οποίοι γίνονται ακόμα και υπεύθυνοι για τη δημόσια ασφάλεια στις περιοχές που ζουν. Αντιλαμβάνεστε πόσο, ε, ε, πόσο άσχημα αισθάνονται, τι αίσθημα ματέως αισθάνονται. Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά ότι η σύγκρουση αυτή ξεπερνάει τα σύνορα της λαϊκής δημοκρατίας του Κόγκο. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν επικοδομητικός διάλογος, διάλογος διαπεριφερειακός με ηγέτες οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στην ειρήνη. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Οι ένοπλες δυνάμεις επίσης και αυτές πρέπει να τις συζητήσουμε γιατί διαρωτώμεθα αν έχουν ε, διερευνηθεί όλες οι δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί στο FDL ένα τελεσίγραφο. Εμείς όμως ως ε, πολίτες διερωτώμεθα αν έχει η διεθνής ε, κοινότητα διαρευνήσει κάθε πιθανή δυνατότητα άσκησης πίεσης πριν φτάσει στη χρήση της βίας. Γιατί με τη χρήση της βίας τις παράπλευρες απώλειες, τις παράπλευρες ζημίες τις ε, επιβαρύνεται ο τοπικός πληθυσμός. Αυτός ο λαός που 20 χρόνια τώρα περιμένει την ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε με δίψα και πείνα αυτή τη μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση του νόμου για τη δημόσια ασφάλεια, ενό νόμου που εγκρίθηκε μένα από το Κοινοβούλιο αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Και άρα η μορφή του συστήματος για την επιβολή της δημόσιας τάξης δεν μας καθησυχάζει. Αν δεν υπάρξει ρύθμιση και εφταξία στους τάξεις της αστυνομίας και του στρατού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Θα θέλαμε να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών στην υλοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο, πλαισίου, ώστε να παρακολουθεί, να επιτηρεί ούτως η ε, τα πράγματα και να διαπιστώνει αν κάτι δεν λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί. Τώρα είναι πολύ ισχνή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και εν τέλει η ενίσχυση της ε, δημοκρατικής διακυβέρνησης και ο σεβασμός του συντάγματος θα πρέπει να βοηθήσουν, μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Μουκβέγκε. Δίνω το λόγο στον κύριο Λουί Μισελ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητέ δόκτωρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ε, η Μαργκρίτ Γιουρσενάρ έχει γράψει μια πολύ ωραία φράση που λέει το εξής ε, το απίθμενο μυστήριο του σύμπαντος ε, τοποθετεί σε τακτά χρονικά διαστήματα πάνω στη γραμμή του χρόνου γενναιόδωρους στυλοβάτες που φωτίζουν τον κόσμο όταν χάνει το δρόμο του. Αυτά είπε η Μαργκρέτ Γιουρσενάρ. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ευτυχής που βλέπω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποτελεί αντιχείο των δικαιωμάτων του ανθρώπου εσάς εδώ δόκτωρα για να χαιρετήσουμε την αξία σας, για να τιμήσουμε το αξιοθαύμα στο έργο σας, το αστήρευτο πνεύμα αλληλεγγύη σας, την αφοσίωσή σας, την δύναμη του χαρακτήρα σας που τολμάτε να καταγγείλετε το ακατονόμαστο, το αβάσταχτο, την ανάγκη ανθρωπιάς, τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται στα βουνά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Με την ακαταπώνητη δράση σας, ε, την επιμονή σας, τη δίψα για την αγάπη των πλησίων, μας δίνεται ένα μάθημα ανθρωπιάς, ε, ε, μετριοφροσύνης και ζωής. Η απλότητά σας, η φροντίδα σας για τον συνάνθρωπο σώζουν τους αδιάφορους όλους εμάς πολλές φορές ε, από την ατίμωση και εξασφαλίζουν στην, μια επίφαση αξιοπρέπεια στη συνείδησή μας. Ε, είσαστε μία από τις πιο όμορφες και τις μεγαλύτερες συνειδήσεις του, όλων των εποχών. Πιστεύω ότι τίποτα δεν, έχουν, δεν, τίποτα δεν έχει χαθεί όσο παραδείγματα όπως το δικό σας ε, δίνουν, ζωή και βοηθούν, ε, δίνουν φωνή στους αδύναμους, τους αφανείς και τους άφωνους. Ε, έχετε κάνει στο Πάντζι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νοσοκομείο. Έχετε δημιουργήσει μια κοινότητα, μια οικογένεια, ένα κέντρο αλληλεγγύης, σεβασμού και δικαιοσύνης. Ε, πρόκειται για ένα ναό που ακτινοβολεί σε όλη την ανθρωπότητα. Ε, μέσω της δράσης σας βοηθάτε να μην επιστρέψουμε σε τέτοιους είδους ε, βάρβαρες πρακτικές, πολεμικές πρακτικές του 21ου αιώνα. Σας έχω ακούσει επανειλημμένως τον τελευταίο καιρό και θα έλεγα ότι η δράση σας ε, είναι μια δράση και μια πράξη αντίστασης. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά την επίμονη στράτευσή σας ε, που έχει ως στόχο να τεθεί τέλος σε αυτές τις βάρβαρες ε, πρακτικές ε, και το έχετε πει επανειλημμένως ότι η δράση σας είναι δράση εναντίον της ατιμορρησίας η, επανηφαίνεται αυτή την υπαρξιακή πεποίθηση ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια ιστορία, στον ίδιο λαό, στην ίδια κουλτούρα, στον ίδιο πολιτισμό. Είσαστε μια γνήσια και τεράστια οικουμενική ε, μορφή που τιμά την Αφρική και όλο τον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας τιμά και σας λέει ότι είναι δίπλα σας σε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχουν οι συνάδελφοι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και είμαι σίγουρη βέβαια ότι θα θέλετε να ακούσετε και μια απάντηση από τον κύριο Μαγκουέγγε. κύριο Πρέντα, Παντζέρη, Τανόκ, Σεβίτσιους, Λόζινγκ και Λογμπίλερ. Αυτοί είναι οι ομιλητές που έχω και ο κύριος Μπασία. η κυρία Χιμένες. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μαγκουέγγε, καταρχάς να σας συγχαρώ για τη βράβευσή σας με το βραβείο Ζαχάροφ 2014. Ήταν πολύ δύσκολη φέτος η επιλογή για μας, διότι ε, οι τρεις τελικοί υποψήφοι τους οποίους έπρεπε να αξιολογήσουμε και για τους οποίους έπρεπε να ψηφίσουμε. Ήταν τρεις υποψήφοι που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Καταρχάς, ήσταν εσείς με τον αγώνα κατά το, της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Είχαμε όμως επίσης και το κίνημα Γερομαϊντάν στην Ουκρανία, καθώς επίσης και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν μέσω της δράσης της κυρίας Λέιλα Γιουνούς. Είμαστε λοιπόν υπέρ και των τριών αυτών σημαντικών δράσεων. Επιλέξαμε εσά κύριε Μαγκουέγγε. Ξέρουμε ότι εδώ και 16 χρόνια προσπαθείτε να βοηθήσετε τι γυναίκε αυτέ οι οποίε ε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τι ιδεχθεί αυτέ πράξει. Χαιρετίζουμε και το θάρρο σα για να συνεχίσετε τον αγώνα σε αυτόν, μολονότι πολλέ φορέ διακινδυνεύετε ακόμα και την ίδια τη ζωή σα, όπω άλλωστε είδαμε το 2012. Συντοποιούμε, όμω επίση ότι εκατοντάδε χιλιάδε γυναίκε υποφέρουν στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, είναι θύματα βιασμών, σεξουαλική βία και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπερασπίσουμε την κάθε μία από τις γυναίκες αυτές, οι οποίες πλήττονται από αυτό το νέο όπλο πολέμου, το οποίο και εσείς αναφέρατε. Θα θέλαμε όμως και μέσω του βραβείου αυτού να προωθήσουμε το έργο όλων εκείνων των ιατρών, που σε αντίξωες συνθήκες προσπαθούν να τιμήσουν τον όρκο του Ιπποκράτη. Τρει είναι οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ οι οποίε συμμετέχουν ε, στη σημερινή συζήτηση και πραγματικά πρέπει να σα πω ότι και για τι τρει αυτέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ το ζήτημα τη βία κατά των γυναικών είναι κάτι που μα απασχολεί πάρα πολύ. Όσον αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, συζητήσαμε ε, διάφορα ζητήματα που άπτονται τη χώρα αυτή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και είπαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να συνεχίσει η χώρα αυτή να είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των βιασμών. Θεωρήσαμε επίση ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην ατιμορρησία όλων των αυτουργών των πράξεων αυτών. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίσουμε από εσά ποιε είναι οι προτεραιότητες οι οποίες εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δώσουμε ένα τέλος στη μάστιγα αυτή την οποία περιγράψατε. Καταδικάζουμε προφανώς όλες αυτές τις πράξεις σεξουαλικής βίας, αλλά θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να τερματίσουμε τις πράξεις αυτές μόνο αν καταφέρουμε τελικά να βγούμε από αυτό το εμπόλεμο περιβάλλον το οποίο πλήττει τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Θα πρέπει λοιπόν να ελοποιηθούν οι συμφωνίες ειρήνευσης οι οποίες ε, υπεγράφησαν στο παρελθόν και θα πρέπει επίσης να αναλάβουν πιο ενεργή δράση οι αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίε ουσιαστικά έχουν ε, εντοπίσει ως βασικό παράγοντα αστάθεια στη χώρα το γεγονός ότι δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις κυβέρνησης και πολλές φορές δεν τηρείται καν το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Εσείς στο παρελθόν είχατε τοποθετηθεί όσον αφορά το ζήτημα της συνταγματικής μεταρρύθμισης στη χώρα σας και θα ήθελα για άλλη μια φορά να μας πείτε ποια είναι η τοποθέτησή σας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Παντσέρη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Μακουέγγε. Θα ήθελα να σας πω ότι φέτος εορτάζουμε την 15η επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας υπαριθμών 1325. Και θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πραγματικά που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Στο ψήφισμα αυτό τονίζουμε τη σημασία του ρόλου των γυναικών όσον αφορά την πρόληψη και την επίλυση των διενέξεων. Και εκφράζονται και κάποιες ανησυχίες ε, για όλους τους αμάχους και για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα πλαίσια τέτοιων ε, διενέξεων, αλλά αναφερόμαστε επίσης και διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά το φύλλο. Η παραβίαση λοιπόν των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ε, κατά τη διάρκεια των ε, διενέξεων αυτών που είχαμε τελευταία χρόνια παραβιάζονται τα δικαιώματα περίπου 40 γυναικών σε καθημερινή βάση και προφανώς εμείς δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοια κατάσταση όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των γυναικών. Μετά την έγκριση λοιπόν του σχετικού αυτού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών 1320 και 1820 και 1325 θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα τελικά ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών να ορίσει ειδικό απεσταλμένο στον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στις εμπόλεμες αυτές διενέξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα πρέπει να υποστηρίξει τα Ηνωμένα Έθνη στο έργο του αυτού και θα ήθελα να γνωρίσω και ποια είναι η δική σας η άποψη όσον αφορά το έργο των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι η αναγνώριση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περνά μέσα από την βράβευση με το βραβείο Ζαχάροφ ουσιαστικά μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε περαιτέρω ένα από τα βασικά ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε μιλάμε για τον Κονγκό, είτε μιλάμε γενικότερα για την Αφρική. Σεβασμός για τα δικαιώματα των γυναικών. Ξέρετε ότι δεν έχουμε μόνο τα θύματα στα πλαίσια των πολέμων, αλλά έχουμε και θύματα τα οποία, τα, τα οποία μπορεί να μην χάουν τη ζωή τους, αλλά παρόλα αυτά στιγματίζονται ανεξίτηλα από τις πράξεις αυτές τις οποίες αναφέρατε εσείς στην παρέμβασή σας. Πράξεις οι οποίες πραγματικά υποτιμούν εντελώς, εξευτελίζουν τις γυναίκες, καταστρέφουν ακόμα και το, το σώμα τους. Θα ήθελα λοιπόν να αφαιρθείτε περισσότερο κι εσείς στο έργο σας, στο έργο που έχετε κάνει ως γυναικολόγος, στο έργο το οποίο κάνετε προκειμένου να αποκαταστήσετε τα γενετικά όργανα των γυναικών και νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδεχομένω θα μπορούσατε να τον απτύξετε λίγο περισσότερο. Είπατε ότι πέρα από τι σωματικέ αυτέ παρεμβάσει συνεργάζεστε και με μια ομάδα ψυχολόγων προκειμένου να βοηθήσετε ψυχολογικά τι γυναίκε αυτέ. Θεωρώ ότι το έργο αυτό το οποίο επιτελείται, η ολιστική αυτή προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι για αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να δώσουμε σε εσά το βραβείο Ζαχάροφ. Μέσω του βραβείου λοιπόν αυτού, τιμώντα εσά, πιστεύω ότι θα πρέπει να τιμήσουμε ακόμα περισσότερο ανθρώπου σαν και εσά που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και που προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο και που λειτουργούν κατά όλων αυτών των διενέξεων που πλήττουν τον πλανήτη μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση αυτή που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Το λόγο έχει ο κύριο Στάνοκ. Πρόεδρε, εδώ είμαι. Εδώ, δόκτωρα Μακουέγκε. Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρου της ομάδας μου που είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου ECR αλλά και ως ε, γιατρός. Είμαι ψυχίατρος συνταξιδοτημένος ε, αλλά ψυχίατρος. Γνωρίζω τις ε, ε, ψυχολογικές και όχι μόνο σωματικές συνέπειες όλων αυτών των πράξεων τις ε, οποίες ε, προσπαθείτε να διορθώσετε. Ε, ενδιαφέρομαι για τη διαδικασία του Κίμπερλι εδώ και πολύ καιρό. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σκέλος των διαμαντιών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε να επεκταθεί και σε άλλου τύπου ορυκτά του, της του Κονγκό αυτή η διαδικασία. Πέρσι φιλοξένησα ένα μικρό σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα ε, της ε, και των βιασμών ως όπλου ε, στην Λαϊκή ε, Δημοκρατία του Κονγκό και μάλιστα συνδεθήκαμε με βίντεο και με το Κονγκό. Όμως ε, ο Βίλιαμ Χέικ από το κόμμα μου ε, φιλοξένησε στο Λονδίνο ένα συνέδριο φέτος για αυτό ακριβώ το ίδιο θέμα ε, και κυρίως εστιασμένο στην Αφρική και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Ε, η βράβευσή σας με το βραβείο Ζαχάρου 2014 για το ζωτική σημασία σε έργο σας είναι μια βράβεση που σηματοδοτεί την ε, σημασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα δεκάδων χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών όχι μόνο στη δική σας χώρα αλλά και σε άλλες ε, σε περιοχές που βρίσκονται σε σύραξη, πολεμική σύραξη. Για παράδειγμα, το πρόβλημα στο Ιράκ και τη Συρία με τον Ισλαμικό στρατό ε, και τα προβλήματα ε, των μειονοτήτων γυναικών οι οποίες όχι μόνο βιάζονται αλλά και πολλούνται ως σκλάβες. Μπράβο λοιπόν, συγχαρητήρια στον Δόκτωρα Μακβέγκε. Το αξίζει το βραβείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάνακο, κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεκούγκε. Συγχαρητήρια όλη η ομάδα μας, ε, Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, είναι στο πλευρό σας. Αξίζετε πράγματι την αναγνώριση και το βραβείο αυτό. Έχετε πλέον το καθεστώς ενός διεθνώς αναγνωρισμένου ανθρώπου, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά στη χώρα σας. Αυτές οι προσωπικές τραγωδίες και οι βαθύτατες πολλές φορές σωματικές πληγές που αφήνουν πίσω τους οι ομαδικοί βιασμοί εις βάρος γυναικών, παιδιών και άλλων δεν πρέπει να μείνουν κρυμμένοι στη σιωπή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα το δημόσιο, το δημόσιο διάλογο για την σεξουαλική βία και κυρίως τη χρήση του βιασμού ως όπλου σε ένοπλες ε, συνθήκες και κυρίως στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Εσείς μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Βλέπετε κάποια τάση να διαγράφεται στη χώρα σας σε σχέση με αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα. Και επίσης, ε, δ. Μουκουέγγε, είναι σημειολογικά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια χρονιά όπου η Ευρώπη εορτάζεται 100 χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 είναι μεγάλος συμβολισμό συμβολισμός της βράβευσης ε, της δικής σας γιατί ταυτόχρονα δίνουμε ένα μήνυμα ότι κάθε πόλεμος, κάθε ένοπλη σύγκρουση παραμένει γεγονός απαράδεκτο και καταστροφικός παράγων. Ο Θεός ευλογεί λοιπόν Ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσετε το έργο σας. Πολλοί ακόμη θέλουν να λάβουν το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το, στο δόκτωρα μου το λόγο για να απαντήσει και θα συνεχίσουμε μετά. Σας ευχαριστώ πολύ Μία ακόμα φορά ζητώ συγγνώμη από την πρόεδρο του πάνελ. Είπα ότι είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών παθήσεων είναι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πρώτη ερώτηση έχει σχέση με την ατιμορρησία. Δεν πρόκειται για την πλειοψηφία των περιπτώσεων και υπάρχει και μια άλλη μικρή μειοψηφία. Η, το, η αίσθηση που εμείς έχουμε και, έχουν και τα θύματα είναι ότι ε, δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόθεση να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της ατιμορρησίας. Ε, επιτρέψαμε στην ατιμορρυσία να εγκατασταθεί και αυτό οδήγησε στην διαιώνιση του φαινομένου, ακόμα και σήμερα. Ο αγώνας κατά της ατιμορρησίας, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να τεθεί στο κέντρο της διαδικασίας καταπολέμησης αγώνα εναντίον αυτών των εγκλημάτων τα οποία αρνούνται την ανθρώπινη φύση του άλλου. Δεν θα πρέπει να σταθούμε αδιάφοροι. Και αν πιστεύουμε, και εδώ πιστεύουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία που έχουμε της ε, μεταβατικής δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το χρόνο, αλλά δεν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα της ατιμορρησίας αν δεν διαθέτει η χώρα τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί οι ξένοι στρατοί βρέθηκαν στο Κονγκό κατά τη διάρκεια μιας μακράς ε, περίοδου. Αυτοί οι στρατοί διέπραξαν σοβαρές παραβάσεις ε, και είναι δύσκολο χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί μια εθνική δικαιοσύνη θα ήταν δύσκολο να απονείμει δικαιοσύνη δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις ομάδες δεν βρίσκονται πλέον στο Κονγκό. Οπότε θα πρέπει να διωχθούν ποινικά οι ε, υπέτη ε, για όλες τις παραβάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερως για τις σεξουαλικές επιθέσεις ε, και υπάρχει η δυνατότητα να διωχθούν ε, και, για, και είναι απαραίτητο και για παιδαγωγικούς λόγους. Στον, στρατό δυστυχώς ε, δεν γινόταν ποτέ φιλτράρισμα ε, αυτών που γινόντουσαν δεκτοί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και γι' αυτό το λόγο πολλοί από τους ε, στρατιώτες ή πολλοί από τους στρατιώτες είναι αυτοί οι οποίοι ήταν υπέτοι για αυτά τα εγκλήματα και μάλιστα πήραν και προαγωγές. Δεν έχει εξηγιανθεί ο δημόσιος βίος ούτε ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό δυσκολεύει πολύ περισσότερο την κατάσταση γιατί θα ήταν σαν να ε, ζητάμε από το θύμα να ζητήσει προστασία από αυτόν ο οποίος κατά βάση τη βίασε το βίασε, το θύμα Για, και τι θα, γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση ε, ε, ο υπέτειος ε, θα απειλούσε μία ακόμα φορά το θύμα ότι κανένας δεν μπορεί να το πειράξει και ότι δεν μπορεί να του κάνει τίποτα κλπ. Συνεπώς πρέπει να γίνει καθάριση στο στρατό και στην αστυνομία. Δεν είναι αργά. Πώς είναι δυνατόν ο λαός να εμπιστευτεί ένα άτομο ε, το οποίο την προηγούμενη ε, μέρα ε, ήταν ο και σήμερα προβάλλεται ως προστάτης. Ε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει στο στρατό στα 10-12 χρόνια τους και κάποια στιγμή ε, μεγάλωσαν, ε, εκδιώθηκαν ενδεχομένω ε, από το στρατό, αλλά ποτέ δεν ε, τους φρόντισαν ψυχολογικά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν παιδιά όταν στρατολογήθηκαν ε, και η ψυχική τους υγεία έχει πληγεί από όλη αυτή την περίοδο. Συνεπώς η μεταβατική δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί σωστά. Δεν υπάρχουν προγράμματα επιδιόρθωσης, δεν υπάρχουν προγράμματα ε, ε, ε ψυχολογικής ενίσχυσης και υποστήριξης και δεν έχει γίνει η μελέτη για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα θύματα των βιασμών και της σεξουαλικής βίας. Εμείς ε, πλησιάσαμε την κυβέρνηση, υπήρχαν ανθρωπιστικές οργανώσεις που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη και η κυβέρνηση δεν την έχει αναλάβει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ε, Επιτροπή Συμφιλίωσης και Αλήθειας ε, ήταν η μόνη πρακτικά επιτροπή που δεν λειτουργήσε καθόλου από όλες όσες δημιουργήθηκαν στη μεταβατική, στη μεταβατική περίοδο. Παρόλο ότι έχουμε τόσα πολλά θύματα, δεν θα έπρεπε να μπορούμε να πούμε την αλήθεια και για αυτά τα θύματα. Δεν θα πρέπει να πούμε ότι αυτό ήταν μια ανοησία που δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Υπήρχε αυτή η ευκαιρία να δοθεί φωνή στα θύματα, να πούν αυτά τα οποία αισθάνονται. Εμείς στο νοσοκομείο το καταφέρνουμε αυτό, γιατί εκεί πολλά θύματα καταφέρνουν να βγάλουν το μίσος τους, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το μοναδικό σημείο που γίνεται αυτό το δικό μας νοσοκομείο. Και θα έπρεπε η κοινότητα να ζητήσει συγγνώμη που δεν κατάφερε να προστατεύσει αυτά τα θύματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε την επανάληψη αυτών των εγκλημάτων. Τώρα, για το θέμα της ε, μεταρρύθμισης του συντάγματος, συνταγματικής μεταρρύθμισης. Πρόκειται για ένα, μια συζήτηση, ένα δημόσιο διάλογο, ο οποίος ε, από ό,τι φαίνεται έχει συρρυκνωθεί. Ενδεχομένως εξαιτίας αυτών που έχουν συμβεί στην Πορκίνα Φάσο. Όμως καλούμε τον ε, πληθυσμό να παραμείνει σε εγρήγορση, διότι αν γίνει συνταγματική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, για να διατηρηθούν ε, οι θεσμοί ε, και τα άτομα ενάντια στην λαϊκή βούληση, τότε μπορεί να οδηγηθούμε ξανά στην εκκίνηση. Θα ήταν κρίμα γιατί θα οδηγούμαστε σε ακόμα περισσότερους θανάτους σε μια χώρα που ήδη έχει υποφέρει πολύ. Καλό λοιπόν τις ε, αρχές να επιδείξουν πολιτική ευθύνη, πολιτική υπευθυνότητα, γιατί ο λαός ζητά να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Η αλλαγή του συντάγματος σήμερα θα μας οδηγούσε να οπισθοδρομήσουμε, να οπισθοχωρήσουμε 10-20 χρόνια. Θα ήταν κρίμα. Αυτό, θα, αυτό έχει ήδη συμβεί στην Πουρκίνα Φάσο και είδαμε τα αποτελέσματα, είδαμε τις συνέπειες. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες εκλογές με το ίδιο σύνταγμα για τρίτη φορά. Ήδη έχει γίνει, έχουν γίνει εκλογές δύο φορές με το ίδιο σύνταγμα. Γιατί να μην αλλάξει το σύνταγμα η επόμενη Βουλή. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ναι, ψυχολογική φροντίδα. Εμείς ξεκινάμε από τη βάση ότι είναι απαραίτητη μια ολιστική αντιμετώπιση. Γιατί αυτό που φέρνει τις γυναίκες στο νοσοκομείο στο Παντζή είναι τα τραύματά τους, τα σωματικά τραύματά τους. Όμως είδαμε ότι η φροντίδα αυτών των τραυμάτων, η νοσηλεία, μόνο σε σωματικό επίπεδο ε, δεν κάνει καλά τις γυναίκες. Ε, οπότε αρχικά ήμουν χειρουργός, αλλά ε, χρειάστηκε να αρχίσω να ακούω τους ασθενείς μου, τις ασθενείς μου και όταν άρχισα να τις ακούω ε, ε, άρχισα να συνδέομαι μαζί τους ε, και διαπίστωσα ότι αυτό δυσκολεύει το ρόλο μου ως χειρουργού. Με εντυπωσίασε η κατάσταση αυτών των γυναικών μια... και ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσω να παίζω και τους δύο ρόλους. Οπότε χρειάστηκα να εγκαθιδρύσουμε και τον θεσμό της ψυχικής στήριξης, της ψυχολογικής στήριξης, συγγνώμη, ε, που παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι ε, η νοσηλεία γιατί για πολλές από αυτές τις ε, γυναίκες χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να γίνουν καλά τα ψυχικά τους τραύματα. Και ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι προϊόντα αυτών των βιασμών. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες έχουν χάσει τις οικογένειές τους, γίνονται σκλάβες, και μένουν έγκυες από ένα βιασμό ο οποίος τις αφήνει με ένα παιδί που είναι το προϊόν αυτής της βίας πράξης. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ε, η φροντίδα αυτών των γυναικών. Και ε, ε, οι γυναίκες ε, αυτές έχουν την τάση να ξαναζούν τα προβλήματά τους ακόμα και όταν φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί η κατάστασή τους. Υποτροπιάζουν. Ε, πρέπει πάντως η ψυχική υγεία να ενταχθεί ε, στις ε, πρωτογενείς φροντίδες, στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας στο σύστημα υγείας της χώρας μου. Μιλήσατε για το Κίμπερλεϊ, για τη διαδικασία του Κίμπερλεϊ και για το θέμα του, του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστο, το μείζον πρόβλημα στη χώρα μου. Δεν μιλάμε για διαμάντια στο Κόγκο. Δεν μιλάμε μόνο για διαμάντια τουλάχιστον. Ε, είμαστε σε μια από περιοχές του κόσμου, αλλά βλέπετε ταυτόχρονα και το πιο φτωχό πληθυσμό του, της Ιφιλίου. Οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ε, φροντίδες υγείας. Έχουμε μεγάλη ε, θνησιμότητα νεογνών. Αλλά ακόμα και όταν φτάνουν, έχουν πρόβλημα σε κάποιες δομές υγείας, αυτές οι δομές ε, είναι αδύναμες. Υπάρχει θνησιμότητα, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν θνησιμότητα 2 ως 3 στις 100.000, σε εμά είναι πάνω από 1.000 στις 100.000 ε, το συγκεκριμένο ποσοστό, είναι τεράστια η διαφορά και προφανώς οι συγκρούσεις για τον ορυκτό πλούτο ε, είναι αποφασιστική σημασίας παράγων, θα θέλαμε πράγματι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ότι θα ψηφίσετε κάποιο νόμο πολύ σύντομα θα θέλαμε αυτός ο νόμος να είναι πολύ πιο περιοριστικός, πολύ πιο αυστηρός, έτσι ώστε ο έλεγχος των ορυκτών να μην γίνεται μόνο στην Ευρώπη, αλλά και επιτόπου, ε, ε, δηλαδή στο σημείο από το, στο οποίο παράγεται. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για να λύσουμε όχι μόνο το πρόβλημα της κρίσης του Κονγκό, αλλά και ε, για να ενταχθεί η προβληματική των δικαιωμάτων του ανθρώπου ε, σε όλη την οικονομική και χρηματοοικονομική σφαίρα δραστηριοτήτων. Πολύ συχνά ε, καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία, των οποίων δεν γνωρίζουμε την προέλευση. Είναι σαφές ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, αρκεί ε, οι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα ορυκτά να ακολουθούν μια στρατηγική που θα υποχρεώνει αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο να μην χρησιμοποιούν τη μεθόδους που δεν πρέπει να χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Βρετανό Ευρωβουλευτή ο οποίος μίλησε για, για την πρωτοβουλία του William Hague ε, που συγκάλεσε 150 χώρες προκειμένου να ε, προβληματιστούμε όλοι μαζί για την ε, στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθεί κατά της χρήσης των βιασμών ως πολεμικού όπλου. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να εμπνεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος ε, τρόπος ε, ε, για να οδηγηθούν οι χώρες να πούνε όχι σε τέτοιες πρακτικές. Πρακτικές οι οποίες επεκτείνονται και διευρύνονται. Ιράκ, Συρία, μιλήσατε για αυτές τις χώρες. υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κομπάζουν ότι πούλησαν 200 κορίτσια ως σκλάβες. Ε, είναι απίστευτο να ακούμε τέτοιου τύπου προτοποθετήσεις, τέτοιου τύπου κουβέντες, τι ε, ε, χαρακτήρα, έχουν τι προσωπικότητες είναι αυτές ο κόσμος θα πρέπει ε, ε, ο κόσμος να βάλει μια κόκκινη γραμμή στα βιολογικά όπλα, στα χημικά όπλα και στη χρήση των βιασμών ως ε, πολεμικού όπλου δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να σιωπούμε και έναντι αυτού του όπλου τώρα υπάρχουν θετικές εξελίξεις στη χώρα μου ε, εξακολουθούμε να ελπίζουμε Χρειάζεται μία μικρή όθηση, ε, ένας πινθύρας έτσι ώστε τα πράγματα να αλλάξουν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ε, στρουθοκαμιλίζει. Αρνείται ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Ε, υπήρχε καταρχήν η ε, η υπόσχεση είναι ότι θα δημιουργηθούν ε, μεικτά δικαστήρια. Ε, εμείς το χαιρετήσαμε ως ε, ανακοίνωση, ως εξαγγελία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα στην πράξη. Αν η κυβέρνηση παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα το πρόβλημα αυτό να λυθεί. Η κατάσταση να βελτιωθεί. Και πιστεύω στη δράση των γυναικών και δεν το λέω επειδή τις φροντίζω, επειδή τις νοσηλεύω, αλλά βλέποντας τι υποφέρουν, πόσο βασανίζονται και βλέποντας τις, την ικανότητά τους να ανασυγκροτήσουν τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους με λίγα μέσα, ε, βλέπω ότι διαπιστώνω ότι η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κάθομαι εδώ στα αριστερά σας. Αξιότιμε κύριε Μουκβέγγε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι υπερηφάνεια που είστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να σας καλωσορίσω εκ μέρους της ομάδας μου της Ενωτικής Αριστεράς της Ευρώπης. Το βραβείο Ζαχάροφ πολλές φορές αξιοποιείται για πολιτικές σκοπιμότητες δυστυχώς. Και γι' αυτό η ομάδα μου συχνά διατυπώνει πολύ επικριτικές θέσεις εναντί των ε, επιλεγέντων για το βραβείο. Χαίρομαι γι' αυτό ακόμη περισσότερο που επιλέγετε εσείς εφέτος για το βραβείο Ζαχάροφ. Ιδιαίτερα θέλω να σας συγχαρώ όπως και οι άλλοι συναδελφοί για την ε, πολύ σπουδαία δουλειά σας. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Θα αναφέρω μόνο ότι και εγώ εργάστηκα σε δημόσια υπηρεσία επί 20 χρόνια, δημόσια υπηρεσία η οποία προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια και είχα τη δυνατότητα άμεσα να γνωρίσω ανθρώπους που ε, στιγματίζονται και σημαδεύονται σε όλη τους τη ζωή από την βία και τη σεξουαλική βία. Όχι μόνο γυναίκες και παιδιά, αλλά και άνδρες και νέα, νέα γόρια, που έφευγαν από εμπόλεμες περιοχές. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όχι μόνο για τα ίδια τα θύματα, αλλά και για αυτούς που τους υποστηρίζουν. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά και γι' αυτό σας οφείλουμε μεγάλη αναγνώριση. Ιδιαίτερα ξέρω ότι η βία εις βάρος των γυναικών δεν είναι χαρακτηριστική σε κάποιο μέρος μόνο του κόσμου. Δεν εμφανίζεται μόνο σε ένα μέρος του κόσμου. Είχαμε και στην Ευρώπη ως μέρος των πολέμων μαζικούς βιασμούς βάρος των γυναικών. Ο βιασμός έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Αναφέρθηκαν νωρίτερα οι στο Ιράκ και τη Συρία αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν 200 οι γυναίκες. Χιλιάδες γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες έπεσαν θύματα απαγωγής, βιασμών, πρώτα για να απολυθούν στη συνέχεια ως σκλάβες στον 21ο αιώνα. Εμείς εδώ στην Ευρώπη και ως Ευρωβουλευτές οφείλουμε να έχουμε την συνυπευθυνότητα με την απονομή αυτού του βραβείου γιατί εάν είναι κομμάτι του πολέμου η σεξουαλική βία θα πρέπει να καταγγείλουμε όχι μόνο αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής πολέμου αλλά τον πόλεμο εν γέννη ως μέσον άσκησης πολιτικής. Πρέπει να ταχθούμε κατά των πολέμων. Πρέπει επίσης να καταγγείλουμε το γεγονός ότι αυτή η μορφή της βίας έχει χρησιμοποιηθεί στο Κονγκό από μέλη στρατιωτικών μονάδων που έχουν καταρτιστεί και εκπαιδευτεί στην Ευρώπη. Μίλησατε κι εσείς για κυβερνήσεις οι οποίες στρέφονται με τις πράξεις τους και τις επιλογές τους κατά του ίδιου τους του λαού. Για κυβερνήσεις οι οποίες εν μέρη έχουν λάβει την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να μην γίνονται συνυπεύθυνε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τέτοια μορφή βίας όπως έχει συμβεί στο παρελθόν ή να υποστηρίζουν τέτοιου είδους βία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα ζωφερότερα κεφάλαια της, απικιακής, της ιστορίας της απικιοκρατίας. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν και πέραν αυτού για να μιλήσουμε για τη φτώχεια ως αναγνωρισμένη πηγή κάθε βίαιης σύγκρουσης. Η φτώχεια λοιπόν πρέπει να καταπολεμηθεί. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται πολιτική η οποία αποβαίνει εις βάρος ενός μέρους των πολιτών αυτού κόσμου. Ναι, πριν από μένα αφήσατε ε, να μιλήσουν οι άλλοι και τώρα θέλω και εγώ να πω μια-δύο φράσεις ακόμα για να τελειώσω. Πρέπει λοιπόν να ταχθούμε κατά των ε, πωλήσεων όπλων από την Ευρώπη σε άλλα μέρη του κόσμου προκειμένου να υποστηριχθούν στρατηγικοί εταίροι, να εξασφαλιστούν κέρδη και να αξιοποιηθούν ε, με πιο αποτελεσματικό τρόπο εξοπλισμοί θανάτου και φόνου. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που συμβαίνουν εις βάρος των γυναικών στη χώρα σας. Η Πρόεδρος, λυπούμε, αλλά αν μιλάτε παραπάνω από όσο επιτρέπετε... Ναι, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα έπρεπε να το έχετε επισημάνει και στους λοιπούς ομιλητές πριν από μένα. Ναι, αλλά ξέρετε, ο χρόνος τελειώνει. Κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους των Πράσινων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ, για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε, που βοηθάτε τις γυναίκες χωριστά, αλλά και που σε πολιτικό επίπεδο αναζητάτε λύσεις για το πρόβλημα. Απάντησατε νομίζω σε όλες τις περισσότερες από τις ε, επιμέρους ερωτήσεις μου. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πέρυσι θελήσαμε δύο φορές να επισκεφθούμε το Ανατολικό Κονγκό και το νοσοκομείο σας. Λόγω όμως ε, των συνεχιζόμενων ε, βιοπραγιών δεν μπορέσαμε να έρθουμε και γι' αυτό χαιρούμε ακόμη περισσότερο που βλέπουμε εδώ σήμερα. Και επίσης θελήσαμε να αποστείλουμε αποστολή, να δούμε μάλλον ε, αποστολή από γυναίκε τη περιοχή των Μεγαλών Λιμνών στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίε μα μίλησαν και μα είπαν τι συμβαίνει και τι αντιμετωπίζουν όταν πάνε στη φυλακή στην αστυνομία για να καταγγείλουν του βιασμού, ε, ότι δεν υπάρχουν φυλακέ στι οποίε να κρατούνται βιαστέ, αλλά ότι ακόμη και ότι βρίσκονται ίδιες αντιμετωπίε με του βιαστέ, γιατί θεωρούνται υπέτειε ε, από την κοινωνία στην οποία ζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε επίση ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο αγώνα κατά τη ατιμορρησία. πρέπει να, να αντιλαμβάνονται και τα θύματα ότι ο βιαστής προσάγεται στη δικαιοσύνη και τιμωρείται γιατί αυτό είναι μέρος της ε, θεραπείας από την οποία πρέπει να περάσουν. Κάτι όμως το οποίο θέλω να σταθώ είναι η μαζική βιασμή. Οι βιαστές προξενούν, διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα, ταυτόχρονα όμως είναι και η επόμενη γενιά τα θύματα. Πρέπει να μιλήσουμε για τη Λιβερία, όπου 60% των ε, γυναικών της κοινωνίας έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Και γι' αυτό πρέπει να στραφούμε στο πώς θα αντιμετωπίσει την επόμενη γενιά μια κοινωνία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και γι' αυτό ρωτάω εάν εσείς ή κάποιες ομάδες στο Κονγκό στρέφεστε για να τίνετε χείρα ε, ή να ζητήσετε χείρα βοηθείας από άλλες κοινωνίες οι οποίες έχουν περάσει στο παρελθόν από αυτή την ε, φρίκη των μαζικών βιαστών, βιασμών για να ρωτήσετε πώς, μπορούν, πώς μπόρεσαν να διαχειριστούν την ε, υπόθεση αυτή και να φτάσουν στην επόμενη γενιά. Ο κύριος Μπασίρ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον ε, δόκτορα Μακουέγγε για την βραβευσή του με το βραβείο Ζαχάροφ, ένα βραβείο σαφώς που ταξίζει πάρα πολύ για τη δέσμευσή του, για το σκληρό του έργο. Όλοι έχουμε μητέρες, αδελφές, κόρες. Εγώ χθες ήμουνα, είχα την τύχη να μπορώ να κάνω μια βόλτα, να βρίσκομαι μαζί με την μητέρα μου, μαζί με την κόρη μου και δεν θα μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ ότι τα κοντινά μου αυτά πρόσωπα θα μπορούσαν ποτέ να πέσουν θύμα τέτοια βία, όπω ακριβώ όμω συμβαίνει με πάρα πολλέ μητέρε, κόρε, εγγονέ στο Κονγκό. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Τα όσα γίνεται στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, δυστυχώ συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και στο Μιανμάρ, στην Ρουάντα, συμβαίνουν επίση στη Σρι Λάγκα και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά στην παρέμβασή σας, αποτελούν τμήμα μιας ολόκληρης στρατηγικής, διότι μέσω του βιασμού καταστρέφεται, βιάζεται όλη η κοινότητα. Παράλληλα, ομαδικά, μαζικά βιάζονται άμεσα ή έμεσα πάρα πολλοί άνθρωποι. Και η γενικότερη στρατηγική οδηγεί στο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αναγκάζονται τελικά να εγκαταλείψουν τι αιστείε του, να εγκαταλείψουν ολόκληρε περιοχέ. Και αυτό ουσιαστικά αντιστοιχεί σε εθνοκάθαρση. Εμεί Πραγματικά το είδαμε αυτό στην Ευρώπη πριν από δύο δεκαετίες στη Βοσνία. Καθώς λοιπόν αναφέρουμε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και από το παρελθόν. Και δούτε το ερώτημά μου. Είπατε πολύ σωστά ότι όντω θα πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημιέ προ τα θύματα. Όντω ότι πρέπει να κινηθούμε στο δρόμο τη δικαιοσύνη. Και είπατε ότι πρέπει να θέσουμε κόκκινε γραμμέ και συμφωνώ μαζί σα γι' αυτό. Πώ μπορεί όμω να γίνει κάτι τέτοιο, πώ μπορούμε να ελοποιήσουμε στην πράξη τη δικαιοσύνη, Πρέπει να απονείμουμε δικαιοσύνη, πρέπει να αποκαταστήσουμε τις ζημιές των θυμάτων αυτών. Πώς μπορεί αυτό να γίνει στην πράξη. Δύο λεπτά θα έχουμε μόνο ακόμα μαζί μας, δέκα λεπτά με συγχωρείτε θα έχουμε ακόμα μαζί μας τους διερμηνείς, επομένω πρέπει να συντομεύουμε προκειμένου να ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές και να απαντήσει και ο κύριος Μαγκουέγγε. Σας ευχαριστώ πολύ νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που παίρνω το λόγο πρώτη φορά εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να χαιρετήσω πραγματικά το θάρρος το οποίο δείχνετε εσείς στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Με συγκίνησε πάρα πολύ η μαρτυρία σας. Και συνδέεται αυτό και με το έργο μου. Ως σοσιαλίστρια συμμετέχω στην Επιτροπή Υπεράσπισης των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χάρηκα πάρα πολύ κύριε Μαγκουέγγε που αναφερθήκατε στην ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει μεταξύ πολιτικής εξουσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, συνταγματικών δικαιωμάτων και συνταγματικών υποθέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν στην Downing Street στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να προωθήσω μία αναφορά στη χώρα μου αυτή όσον αφορά τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και αναφέρομαι σε γυναίκες οι οποίες έρχονται στο Μένο Βασίλειο για να ζητήσουν άσυλο. Γυναίκες που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από εμπόλεμες διενέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο στη δική μου τη χώρα, αλλά παντού στον κόσμο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές. Και μάλιστα πρόσφατα μάλλον πριν από λίγο μιλούσαμε στην Ολομέλεια για το γενικότερο πλαίσιο όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άκουσα ορισμένους συνάδελφούς μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πέρα που είπανε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να θέσουμε μόνο μία προτεραιότητα όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια, όσον αφορά συγκεκριμένα την εξάλληψη της ελονοσίας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο πόσο σημαντική είναι η βοήθεια την οποία σας δίνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι. Πόσο σημαντική είναι η δική μας η χρηματοδότηση όσον αφορά το έργο το οποίο σας επιτελείτε για να βοηθήσετε τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Πρόστα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο επιτελείτε και θα ήθελα να αναφερθώ στο ακόλουθο. Πάρα πολλά πράγματα ήδη έχουμε πει, πάρα πολλά πράγματα ήδη έχουμε καλύψει μέσω των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Θα ήθελα πάντως και εγώ να πω ότι το πρόβλημα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα συμβαίνει όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, αλλά ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο για παράδειγμα στα Βαλκάνια. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται για ένα νέο πρόβλημα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ανέκαθεν βλέπαμε στο παρελθόν κάθε φορά που διεξάγεται ένας πόλεμος. Μια βία η οποία ασκείται συνεχώς σε περιόδους πολέμου κατά των γυναικών. Αναφερθήκαμε επίσης ε, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερθήκαμε επίσης ε, σε μια, στην απόφασή μας να σας δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ και μας δόθηκε και η δυνατότητα κατά αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς όμως να έχουμε τονίσει δεόντως την πολιτική διάστασή του. Σε αυτό θα θέλω να επιμείνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο την ίδια την κοινωνία των πολιτών παράλληλα με τους ε, πολιτικά ηθήνοντες. Και θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον να βλέπουμε συνεχώς τις επιζήμιες αυτές συνέπειες για τις γυναίκες αυτές οι οποίες πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών αυτών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόστε. Κύριε Μακουαίκη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα αγωνιζόμαστε για να επεκτείνουμε το μοντέλο υποδοχής και μέρημνας του νοσοκομείου Πάντση και σε άλλες περιοχές που γνωρίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τα δικά μας. Είχα επαφές, συνάντησα μια γυναίκα από το Αφγανιστάν, θα ήθελα να το επισημάνω αυτό που ήρθε να μας μιλήσει, γιατί πιστεύει ακράδαντα και μάλιστα όταν της έκανα την παρουσίαση ξέσπασε κλάματα και μου είπε οι γυναίκες στη χώρα μου ζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πούνε, δεν ξέρουν σε ποιον να στραφούν και ζουν μέσα στον πόνο τους, πεθαίνουν μέσα στον πόνο τους και εγώ θα ήθελα αυτό το μοντέλο μου λέει να μπορέσουμε να το εισαγάγουμε στο Αφγανιστάν. Είμαστε σε επαφή με ομάδες στην Πουρκίνα Φάσο, όπου πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε σχέση και με, τις, ε, με τους σεξουαλικούς ακροτηριασμούς, με τους ακροτηριασμούς ε, σεξουαλικών οργάνων ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχέση με τη δουλειά μας. Θα ήθελα να σας πω ότι χωρίς την υποστήριξη του προγράμματος ΕΚΟ δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε, γιατί η ιατρική φροντίδα αλλά και η ψυχολογική φροντίδα στο νοσοκομείο μας καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΚΟ. Βοήθεια για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γιατί έχουμε να κάνουμε με γυναίκες ε, άπορες ουσιαστικά τις οποίες μπορούμε να φροντίσουμε δωρεάν και πλήρως γιατί χωρίς αυτή την υποστήριξη δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Και κλείνοντας θα ήθελα να, περάσω, να αναφερθώ στις κόκκινες γραμμές με τιμά ιδιαίτερα και με κολακεύει που αναφερθήκατε στο ζήτημα αυτό το να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή όπως είπατε ε, σε σχέση με το βιασμό ως ε, όπλο στον πόλεμο είναι ευθύνη για τον καθένα μας είναι ευθύνη για ολόκληρη την κοινότητα Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κοινότητά μας, στην κοινωνία μας, σε συνομιλία με φιλάρχους που στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο ουσιαστικά διατυπώνουν τους κανόνες της κοινωνίας και κέρουν του σεβασμού των πολιτών και βλέπουμε ότι πολλές είναι παραδόσεις οι οποίες απαγορεύουν την αιμομιξία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν ή και καταδικάζουν τον αιμομίκτη, γιατί να μην καταδικάσουν και να καταγγείλουν και το βιασμό. Έτσι μπορούμε να καταστήσουμε κοινά αποδεκτή την καταδίκη αυτής της πρακτικής στην κοινωνία. Επίσης, σε ευρύτερο επίπεδο, όταν εφαρμόζονται, όταν ε, εγκρίνονται νόμοι πρέπει και να υλοποιούνται. Έχουμε έναν από τους καλύτερους, από τα καλύτερα νομοθετήματα στον κόσμο κατά τον βιασμό. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν βοηθάει το θύμα, δεν μπορεί να φτάσει στην απόδοση δικαιοσύνης το θύμα. Πρέπει λοιπόν ο Δήμιος να αντιληφθεί ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται τέτοιου είδους εγκλήματα και ότι είναι υπεύθυνο και υπόλογος. Για τη διεθνή κοινότητα υπάρχουν χώρες γνωστές, ένοπλες ομάδες γνωστές, άτομα γνωστά που τη μέθοδο αυτή την μετέρχονται εις βάρος του, του άμαχου πληθυσμού εις βάρος των γυναικών. Θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες δράσεις, αποτρεπτικές δράσεις, πολύ αποτελεσματικές. Εγώ είπα, μια ομάδα φερρυπίν ένοπλη που χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή ή μια στρατιωτική μονάδα που ανεγνωρισμένα έχει χρησιμοποιήσει μια τέτοια μέθοδο, έστω και αν έχει την προστασία του κράτους τους, θα μπορούσαν εφερειπή να δουν να τους απαγορεύεται η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κράτη, να με τους χορηγείται θεώρηση διαβατηρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί, αναγνωριστεί ως υπέτειος, έστω και ένα χέρι της προστασίας των κρατικών του αρχών, αλλά ξέρουμε ότι έχει διαπράξει βιασμούς ως ε, όπλο πολέμου ή χρησιμοποιεί ε, για λόγους τέτοιου στρατιωτικούς ε, τέτοια εγκλήματα εις βάρος ανθρωπότητας, δεν μπορεί να πατήσει το πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας τρόπος να τους αποθαρρύνουμε. Σας ευχαριστώ. Μπορούν να επιβληθούν να παγώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη περισσότερο παγκόσμιας κοινότητας μπορεί να αναλυφθούν μέτρα αποτρεπτικά που θα υποχρεώσουν ανθρώπου αυτού να αντιληφθούν ότι θα κάτσουν εδώ του κατηγορουμένου ολόκληρη ανθρωπότητα, ολόκληρη διεθνού κοινότητα, εάν διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μα να κάνουμε και να αντιληφθούμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, γιατί τότε και τότε πρέπει εμεί να χαράξουμε όλοι μα και ο καθένα στο επίπεδό του αυτήν την κόκκινη γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί, πόλο δε μάλλον που φτάνουμε πια στη δυνατότητα να συναντιόμαστε και να συζητούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Ακούγοντα Ακούγοντάς σας, ακούγοντας ανθρώπους σαν και εσάς, ο κόσμος γίνεται πιο αποδεκτός. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.